να κάνω μια ανακοίνωση για την εκλογή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια θέση πλέον είναι κενή μετά την εκλογή του κυρίου Ρέν στις εθνικές του εκλογές. Σύμφωνα με το άρθρο 15 πρέπει να προταθούν υποψήφοι. Το EFTD προτείνει τον κύριο Φάμπιο Μάσιο Καστάλτο, η φιλελεύθερη την κυρία Γέτεν Μάκη. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου 12 η ώρα. Ευχαριστώ. θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξή μας. Ε, πρώτα απ' όλα όμω να κάνω και μια ανακοίνωση ε, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με ε, πρόταση για απόφαση η οποία είχε υποβληθεί χθες, είχε περιθώριο